Ψηφίσατε όλοι. La votazione è... Τέλος ψηφοφορίας. La relazione è approvata. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Σόλτ, δεσμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγή ή σημερινού. Πάλι είναι μία μόνη ψηφοφορία, ονομαστική άρχεται ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Τέλος La relazione è approvata. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Ντεπρέ για την κινητοποίηση του περιθωρίου για πρόβλεπτε ανάγκε το 2014. Ολόκληρο το ψήφισμα, ονομαστική ψηφοφορία, έρχεται η ψηφοφορία. Τέλο votazione chiusa. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Έκθεση ΔΕΠΡΕ για το σχέδιο διευθυντικού προϋπολογισμού, το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. La relazione è Εγκρίνεται. Ακόμα ένα ψήφισμα ΤΕΠΡΕ, σχέδιο δοτικού προπολογισμού 4-2014, μία ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνατε. Relazione Sulin sulla mobilitazione Έκθεση Σούλεν για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη, πλημμύρε στην Ιταλία, σημισμοί στην Ελλάδα, χιονοθύελα έλα στην Σλοβενία, πάγο και πλημμύρε στην Κροατία. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. La votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. La relazione è approvata. Εγκρίνεται. Relazione progetto di... Έκθεση ΔΕΠΡΕ, σχέδιο ζωτικού προπολογισμού υπαριθμών 5 2014. Μία ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σχέδιο ΔΕΠΡΕ, σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 6-2014, μία ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φερνάντες, Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη πλημμύρε στη Σερβία, Κροατία και Βουλγαρία. Μία ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, έκθεση ΔΕΠΡΕ για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7-2014, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση ΔΕΠΡΕ. Σχέδιο δοσοτικού προπολογισμού 8-2014. Μία ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ε, της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ντεπρέ Λεβαντόφσκι. Σύστημα ιδίων πόρων τη Ένωση. Προσαρμογέ των εθνικών συνεισφορών των κρατών μελών. Μία ψηφοφορία. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μούρεζαν. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιοχέ που πλήττονται από καταστροφέ. Μία μόνο ψηφοφορία ονομαστική χρειάζεται ειδική πλειοψηφία πάνω από το 1 τρίτο των ε, ψηφισάντων. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione Τέλος ψηφοφορίας. Υπάρχει η ειδική πλειοψηφία και εγκρίνεται η έκθεση Μούριζεν. Έκθεση Γκαρδία Ζαμπάλ Ρουμπιάλ. Κινητοποίηση του μέσου ευελιξία υπέρ των προγραμμάτων των Διευθυντικών Ταμείων για την Κύπρο. Και εδώ χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν. Μία μόνο ψηφοφορία. Άρχεται. Τέλος. Έχουμε την απαραίτητη πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στον προϋπολογισμό του 2015. Θέση του Συμβουλίου, ε, τίτλος 1, τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το, η τροπολογία. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 5 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 6 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 ε, υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε την έκθεση Γκουαρδιαζαμπάλο Ρουμπιάλ Χολμάιερ για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015. Ξεκινάμε παράγραφος 1, τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 μετά από την παράγραφο 14 πρώτο κομμάτι ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15 μετά από την παράγραφο 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 έχει αποσυρθεί. Μετά από την παράγραφο 10, τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 11, τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 12, τροπολογία 21 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Τροπολογία απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 14, η τροπολογία 24, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 15, 23, η, η τροπολογία 23 έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 15, τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. La votazione è Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Μετά από την παράγραφο 16 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο Απορρίπτεται. Η κυρία Ματίας για διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να κάνω μία μικρή διευκρίνηση για το Προεδρείο, γιατί όταν είδα τον κατάλογο της ε, ψηφοφορίας είδα ότι η τροπολογία 30 δεν θεωρηστήκε αποδεκτή για την ψηφοφορία. Θέλω να ρωτήσω γιατί δεν έγινε δεκτή, αφού ήδη είχαμε ψηφίσει τον διορθωτικό προϋπολογισμό του 14. Αυτό που λέω στο 30, που είναι η τροπολογία της ομάδας μας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης τα μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμβάλλουν με το 7% ε, του μισθού μας, του μισθού τους ε, ως ένα ποσοστό αλληλεγγύης για τους λαούς που υποφέρουν, όπως επιβάλαμε και στους υπαλλήλου του Κοινοβουλίου. Αφού έγινε δεκτό για το 2014, γιατί να μην είναι αποδεκτή η τροπολογία αυτή και για φέτος, για τον επόμενο χρόνο. Αυτή η τροπολογία έχει επανειλημμένα υποβληθεί στο παρελθόν και ποτέ δεν έχει γίνει δεκτή. Δεν υπάρχει προηγούμενο λοιπόν. Περνάμε μετά από την παράγραφο 18 στην ε, τροπολογία 31. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορία. Emendamento è respinto. Emendamento 32. Απορρίπτεται 32. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 33. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 20, τροπολογία 34. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μα είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άμα θέλετε όμως ηλεκτρονικό έλεγχο, ας το κάνουμε. Περάστε. La votazione è Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, έχει το λόγο ο κύριος Αρτουής, πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρο για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, διότι είναι πάρα πολύ ε, δύσκολη κατάσταση ε, παρόλα Παρ' όλα αυτά δίνουμε στην Ένωση τον προπολογισμό που χρειάζεται. Θέλω να ευχαριστήσω όλου εκείνου οι οποίοι συνεισέφεραν στο να επιτευχθεί η συμφωνία στον τριμερή διάλογο. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιταλική Προεδρία. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Γεωργίεβα. Ε, τι συζητήτριέ μα, τα μέλη τη Επιτροπή Προπολογισμού και κάθε έναν από εσά ξεχωριστά, αγαπητοί συνάδελφοι. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι ε, εξ ονόματος του εγώ προείδρευσα στην συνδιαλλαγή ε, για τρεις λόγους μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ε, θα αρχίσει από το 2015 ένα σχέδιο εξόφλησης των λογαριασμών στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να διαφυλεχθεί η αξιοπιστία και το κύρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερος λόγος. Περιμένουμε εναγωνίως τον διορθωτικό προϋπολογισμό που θα ανοίξει το δρόμο για το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισεκατομμύριων. Και τέλος, Αναμένουμε ε, τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επίπεδου υπό την ηγεσία του κυρίου Μόντι για τους ιδίους πόρους και η Επιτροπή Προπολογισμών θα φροντίσει κάθε δαπάνη μας να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ε, να είναι η απόδειξη για την ανταγωνιστικότητα και ε, την απασχόληση στην Ευρώπη και καλά Χριστούγεννα. Onorevole Artui, ricambiamo gli και εμεί θέλουμε να παραλάβουμε τι ευχέ για τι γιορτέ. Θέλει να λάβει το λόγο το Συμβούλιο. Grazie, Presidente. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Αντιπρόεδρε Γεωργίευα, κύριε και κύριοι. Σύντομα να πω ότι το Συμβούλιο ε, καταγράφει με ικανοποίηση ότι το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία που επετεύχθη στο τριμερή διάλογο της 8 Δεκεμβρίου 2014 και άρα ο προϋπολογισμός, για τον προϋπολογισμό 2015 καθώς και για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς για το 2014 που τώρα εγκρίνονται επισήμως. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω άλλη μια φορά το πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών, κύριο Αρτουή, την κυρία Γκαρδία Ζαμπάλ, Χολμάγερ και Ντεπρέ, τους εισηγητές ε, για την θετική του στάση στη διάρκεια όλης της δημοσιονομικής διαδικασίας που οδήγησε στο, ε, ε, στην αίσια έκβαση και να σας ευχηθώ επίσης με την ευκαιρία σε όλους καλές γιορτές σε εσάς Πρόεδρε και σε εσάς αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστούμε κύριε Τελαβέντοβα. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε χωρί τροπολογίε στη θέση του Συμβουλίου τη 12η Δεκεμβρίου 2014 όσον αφορά το Γενικό Σχέδιο Προπολογισμού που υποβλήθηκε από την Κομισιόν. Η διαδικασία του προπολογισμού για το 2015 έτσι ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 314 της συνθήκης που ε, διέπει την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλώνουμε ότι ο προϋπολογισμός για το 2015 εγκρίθηκε οριστικός. Περνάμε στο ψήφισμα, πρόταση μάλλον ψηφίσματος για τις ε, οδικές μεταφορές. Μετά από την παράγραφο 3, τροπολογία 1, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Volete il check, ma è stato respinto. Alla votazione aperta. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Απορρίπτεται το κείμενο. Ε, νομίζω ότι το βλέπετε. Μετά την αιτιολογική σκέψη, η τροπολογία 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ συγγνώμη 4 με ναι, ονομαστική κλίση άρχεται πέρας απορρίπτεται τροπολογία 5 πάλι με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μετά την τελευταία σκέψη M, τροπολογία 6 μονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. εποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Χρειάζεται εδώ ειδική πλειοψηφία. La votazione è chiusa. Πέρασε. Εγκρίνεται το ψήφισμα και αποκτά και έχει την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται. Proposta di risoluzione della πρόταση ψηφίσματος Επιτροπής Περιβάλλοντος για την ποιότητα το, της βενζίνης και του διζελ. Χρειάζεται ειδική πλειοψηφία το σύνολο του ψηφίσματος Μορμαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. La votazione è Πέρας ψηφοφορίας. δεν επετεύχθη η ειδική πλειοψηφία. 337 εναντίον 325, αλλά δεν έχει την ειδική πλειοψηφία, δεν εγκρίνεται επομένω. Piano in materia di rigetti nel Mar Baltico, la proposta di risoluzione del gruppo. Απορρίψει στη Βαλτική θάλασσα, ο, o ο κ. Ζομπάτσι, ο συντάκτης της, ε, του ψηφίσματος, θα λάβει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό τροποποιεί την ε, κατεξουσιοδότηση ε, πράξη τροποποιώντας σε 38 εκατοστά και όχι 35 εκατοστά το ελάχιστο μήκος για την προστασία των βακαλάων. Δεν μπορεί κανείς να προστατέψει τα αλλιεύματα με το να μειώσει το ελάχιστο μη, μήκος τους. Εάν καταστρέφετε τα νεαρά ψάρια δεν μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον. Λόγω αυτής της έλλειψης προστασίας έχει μειωθεί ο αριθμός των μπακαλιάρων στην Βαλτική θάλασσα. Θέλετε, η Κομισιόν θέλει να μειώσει το μέγεθος το ελάχιστο, αλλά εγώ ζητώ να υποστήριξετε το ψηφισμά μου. Ευχαριστώ πολύ ψηφίσουμε το σύνολο στο σύνολό του με ονομαστική κλίση. Χρειάζεται και εδώ ειδική πλειοψηφία, άρχεται ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Πέρασε. Απορρίπτεται. Passiamo αλλά Πρόταση ψηφίσματος των πρασίνων σε σχέση με την ασφάλιση και την αντασφάλιση. Χρειάστηκε εδώ ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε το σύνολο με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο ψήφισμα τη Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών για την Ευρωπαϊκή Εσωτερική Στρατηγική Ασφάλεια. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά από την παράφορα 2 τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ψηφί κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο ψήφισμα το κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων για την αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από παλιά υποστηρίκτη μιας άλλη Ισλαμικής χώρας που είναι το Σομάλιλαντ. Στις 3 Σεπτεμβρίου φέτος έγραψα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστειλα μια γραπτή ερώτηση. Μα δεν είναι διαδικαστικό αυτό τώρα. Το 2014 ο πρόεδρος διακόπτει. Κοιτάξτε, δεν είναι διαδικαστικό. Δεν είναι point of order. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες. Πρόταση, κοινή πρόταση ψηφίσματος πέντε ε, πολιτικών. Παρακαλώ καθίστε. Η πρόταση, λοιπόν, η κοινή... Το... Με ονομαστική κλίση. Δεν είναι διαδικαστικό αυτό το οποίο κάνετε. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για τη Σομαλιλάνδη. Έχετε κάνει μια δήλωση αλλά δεν είναι διαδικαστικό θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο σημείο στην μέρες. Σας παρακαλώ να σταματήσετε. Χωρί μικρόφωνο βουλευτής. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να συμφωνούμε για πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι διαδικαστικό θέμα. Για ποιο άρθρο του κανονισμού κάνετε έκκληση, κύριε Πρόεδρε, λέει ο βουλευτή. Χωρί μικρόφωνο. Sento Κοιτάξτε, δόξα ο Θεό ε, καλά, ε, ε, ανάψτε το μικρόφωνο για να σα ακούω καλά. Ναι, είναι σημαντικό το θέμα. Έθεσα γραπτό ερώτημα σε σχέση με μια άλλη μουσουλμανική Ισλαμική χώρα, τη Σομαλία. Μα ακούστε, τη Σομαλιλάνδη, με συγχωρείτε. Ναι, αλλά ακούστε, η Κομισιόν απάντησε στις 4 Οκτωβρίου 2014 και απάντησε ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να αναγνωρίζει κράτη. Μόνο τα μεμονωμένα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό, όπως έχει κάνει η Σουηδία. Εγώ σας ζητώ ως πρόεδρο αυτού του Κοινοβουλίου να μην δώσετε αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα, περνάμε στην ψηφοφορία. Κοινή πρόταση ψηφίσματος πέντε ομάδων. Κοιτάξτε, επειδή όλοι καλά είμαστε, είναι σαφές ότι εδώ δεν έχει σχέση αυτό που είπατε. Έχουμε κοινή πρόταση ψηφίσματος από πέντε ομάδες. Ονομαστική κλίση άρχεται. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Ζήτησε τον λόγο ο κύριος Βέμπερ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ε, όλοι αισθανόμαστε τη σημασία του θέματος αυτός και θα ήθελα να, ε, ε, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους ε, βουλευτές που συνεργάστηκαν. θέλουμε δύο κράτη, ένα Ισραήλ δημοκρατικό, ειρηνικό που να το αναγνωρίζουν όλοι οι Παλαιστίνοι και μια ανεξάρτητη Παλαιστίνη που να αναγνωρίζει και το Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα δηλώσαμε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα πρέπει να είναι το τέλος της διαδικασίας. Δεν πρόκειται ούτε για άμεση ούτε για ανεφόρον αναγνώριση. Είναι η κατάληξη μιας διαδικασίας, η τελική έκβαση, το τελευταίο βήμα. Όσο σημαντικά ε, και αν είναι αυτά όμως ήταν σημαντικό και το σημερινό βήμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόφαση αυτή. Ο κύριος Πιτέλα. Κύριε Πιτέλα, σύντομα παρακαλώ. Ναι, και εγώ πρόεδρε, και εγώ πιστεύω πως πρόκειται για μια ιστορική σημασία μέρα και ότι ολόκληρο το Κοινοβούλιο ε, ε, προέβησε μια σημαντική ψηφοφορία με στόχο να ανοίξουν ελεύθερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις όρους των ε, εξτρεμιστών και των φανατικών, των φανατισμένων. Η ομάδα μου δούλεψε σκληρά, με, με... υπομονή, ισορροπία και με πάθος. Αλλά αυτή είναι νίκη όχι της πολιτικής ομάδας, όχι ενός τμήματος, αλλά ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πρόκειται για τη νίκη της ειρήνης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι η δική μου πολιτική ομάδα εβδομάδες και μήνες ολόκληρους έχει εργαστεί για αυτό το ψήφισμα και αποφασίσαμε προς ε, ε, το όφελος ε, της Παλαιστίνης, του κράτους Παλαιστίνης να υπερψηφίσουμε για την αναγνώριση υπέρ των κρατών παρόλο που έχουμε μεγάλη δυσκολία ε, με τις προϋποθέσεις που τίθενται για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, του Παλαιστινιακού κράτους. Δεν το θεωρούμε σωστό. Θεωρούμε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι η προϋπόθεση για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και όχι το αντίστροφο. Ο κύριος Φερχόφστατ. Ναι, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι συνεργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτό το ψήφισμα που πέρασε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Είναι πάνω από 500 βουλευτές που το υπερψήφισαν. Τώρα δεν πιστεύω ότι είναι η στιγμή να αρχίσουμε να δίνουμε ο καθένα την ατομική του ερμηνεία για το ψήφισμα αυτό. Αυτό που έχει σημασία ποιο είναι. Επιτέλους το Κοινοβούλιο έλαβε θέση και αυτό δίνει ένα σαφές μήνυμα προς τον έξω κόσμο ότι η Ευρώπη επέστρεψε σε αυτό το σημαντικό θέμα. Και δεύτερον, δεύτερον η μεγαλύτερη σημασία ε, και το μεγαλύτερο μήνυμα είναι ότι δίνει σαφή εντολή στην κυρία Μογκερίνη για να προχωρήσει, πράγμα που χρειάζεται οπωσδήποτε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρία Χάρμς, θέλω να πω και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή όσο και αγωνιώδη η διαδικασία ψήφισης μέχρι χτες και αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να πούμε κάτι έστω και συμβολικά σε αυτή την υπόθεση εάν καταφέρουμε αυτό που είπε ο Γκίφερ Χόφστατ ότι η Ευρώπη να επιστρέψει ισχυρή με την κυρία Μογκαρίνη σε αυτή τη σημαντική διαπραγματευτική διαδικασία, τότε δεν βοηθάει η επιστροφή στην παλιά ιδεολογική αντιπαράθεση. Και κύριε Βέμπερ, νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε για αυτά που είπατε εσείς, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες και τις επόμενες εβδομάδες να είναι στοιχημένο, ενωμένο πίσω από την κυρία Μογκερίνη. Κοιτάξτε, δεν θα ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση για το θέμα, δεν ανοίγει συζήτηση για το θέμα. Μόνο επειδή ήταν σημαντική ψηφοφορία έδωσα στους επικεφαλείς των ομάδων, δεν μπορείτε να διακόψετε. Θα πρέπει να περιμένετε να απαντήσω γιατί ζήτησε το λόγο ο κύριος Φάρατς. Επειδή δεν πρόκειται για συζήτηση, δίνω μόνο το λόγο στους επικεφαλείς των ομάδων και μετά θα επανέλθουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι άσχετο το τι πιστεύει ο καθένας από εμά σε σχέση με το θέμα του Ισραηλοπαλαιστιλιακό κύριε Πρόεδρε. Εσείς λέτε ότι είστε κοινοβούλιο και αν είστε κοινοβούλιο, τότε μάλλον πιστεύετε σε κανόνες και στο καράτος δικαίου. Ο συνάδελφος Γκάρντερ τον οποίον φωνάζοντας τον σταματήσατε, με το, οι ίδιοι οι αντιδημοκρατικοί που φωνάζετε και τώρα, κύριε Πρόεδρε, τον αγνοήσατε. Πριν από λίγε εβδομάδε μόλι έγραψε στην Κομισιόν για την αναγνώριση ή όχι της Βρετανικής Σομαλιλάνδης. Του είπαν ότι η οχι τη βρετανικη Σομαλιλάνδη. του ειπαν οτι η κομισιον νησιών δεν έχει τη δυνατότητα, την εξουσία ή το δικαίωμα να αναγνωρίζει νέα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό και το αίτημα σας που σας υπέβαλε αυτό, ότι αυτό το ψήφισμα ήταν ε, απαράδεκτον. Και σας ζητώ το, ρωτώ τώρα να το δείτε και να το αποφασίσετε και να διαγραφεί αυτή η ψηφοφορία, γιατί δεν μπορούμε να λέμε στην κυρία Μογκερίνα να προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από δική τη παραδοχή δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κάλεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου, όπως και πολλές άλλες ομάδες, είχαν μια εσωτερική συζήτηση για τα θέματα αυτά. Πολλοί θεωρούσαν, ανεξάρτητα από την προσωπική τους θέση για την Παλαιστίνη και την αναγνώρισή της, ότι αυτό είναι ένα θέμα για τα κράτη-μέλη και όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει ένα κράτος όπως η Παλαιστίνη. Τώρα έχουμε ψηφίσει όμως και χρειάζεται σαφήνεια. Αν θέλουμε να επιτύχουμε μια βιώσιμη ειρήνη στην Παλαιστίνη, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Θα πρέπει η Φατάχ να αντιμετωπίσει τα θέματα διαφθορά. Η Χαμά θα πρέπει να αποκηρύξει την τρομοκρατία και το Ισραήλ και η κυβέρνηση Νετανιάχου θα πρέπει να σταματήσουν να χαλιναγωγήσουν του επικισμού και να επανέλθουν στα σύνορα του 1967. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε σε βιώσιμη ειρήνη μεταξύ των δύο αυτών παρατάξεων. Κύριε Φάραντ, το κείμενο δεν είναι νομοθετικό. Πρόκειται μόνο για ένα πολιτικό έγγραφο, το οποίο στηρίζει την δράση στην οποία προβαίνουν κάποια κράτη. Οπότε το έγγραφο αυτό ήταν απόλυτα αποδεκτό, παραδεκτό μάλλον. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματο τη ομάδα ΑΛΤΕ για την προστασία των εργαζομένων στις, ε, βιομηχανίε. Ψηφίζουμε στι βιομηχανίε Χάλιβα. Ψηφίζουμε στο σύνολο υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος, στην κοινή πρόταση ψηφίσματο των τριών πολιτικών ομάδων μετά από τον τίτλο την τροπολογία 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 1 υπάρχει τροπολογία, προφορική τροπολογία Νταμάτο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ζητώ από τους συναδέλφους να αφαιρέσουν από την παράγραφο 11 την πόλη του Τάραντο γιατί πρόκειται ε, την ε, πιο Ευρώμικη βιομηχανία της Ευρώπης που εξακολουθεί να παραβιάζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ε, πρόκειται για ε, μια βιομηχανία τελείω μη βιώσιμη, έχει ήδη καταδικαστεί από το, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, είναι υπό εξέλιξη διάφορες ποινικέ καταγγελίες αλλά και διαδικασία κατά παράβαση. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανάκαμψη ολόκληρης της επαρχίας του Τάραντο. Του Τάραντα. Μάλιστα. Ε, υπάρχει κάποιος που είναι αντίθετος στην πρόταση αυτή τροπολογίας. Ναι, 40 βουλευτέ, πάνω από 40 βουλευτέ λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχτούμε την προφορική σα τροπολογία, οπότε ψηφίζουμε σε τρία τμήματα την αρχική τροπολογία. La prima parte. La prima parte. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 38 στην παράγραφο 9 σε δύο τμήματα και τα δύο με ονομαστική κλίση αρχίζει η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Στην παράγραφο 9 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, δεύτερο τμήμα, ε, μάλλον συγγνώμη διορθώνει ο πρόεδρος, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Αρχικό κείμενο. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 12, τροπολογία 40, ονομαστική κλίση, άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 13, τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, παραγραφός 13. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ποιοι είναι υπέρ στο δεύτερο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 16, τροπολογία 5, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17. Το πρωτότυπο κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, Α ελέγξουμε όλα. έχει εγκριθεί. Απέρτα. La votazione è ε, Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παρακαλώ όμως όλοι να ψηφίζετε ή να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να ελέγξω καλά. Παράγραφο 18, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 23, η τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. <laughs> Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Μετά την παράγραφο 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Μετά από την παράγραφο 28, τροπολογία 6, ονομαστική ψηφοφορία. Ποιοι είναι, ε, μάλλον ε, ψηφίστε παρακαλώ. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μετά από την παράγραφο 29, τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εντάξει, έλεγχος. La votazione è chiusa. Εγκρίνεται. Παρακαλώ να ψηφίζετε όλοι γιατί διαφορετικά από εδώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ψηφίζετε. Λοιπόν, 45, ε, ε, μάλλον 18 συγγνώμη, με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Votazione è chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. La Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μετά την πειράγραφο 30, τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Αλλά πολύ δεν σηκώνεται τα χέρια. απέρτα. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Α ελέγξουμε άντε και για τη 17. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 31, Παράγραφος 31, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 μετά την παράγραφο 31. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά την παράγραφο 33 τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 στην παράγραφο 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά από το δεδομένο ότι το, ε, τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά από την αιτιολογική D, τροπολογία, ε, e, ε τροπολογία 12 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 30 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Όχι, υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 31. Ονομαστική κλίση. Τέλος πληροφορίες. Απορρίπτεται. Μετά από την αιτιολογική L, τροπολογία 1, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Για την τροπολογία 1, μετά την αντιλογική σκέψη L, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Αγκρίνεται. Η τροπολογία 14. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 32 Πέρα. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Q. Η τροπολογία υπερθών 33. Ψήφι πέρα Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 στην αιτιολογική σκέψη ΤΑΦ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος τώρα υπέρ κατά αποχές χρειάζεται έλεγχος νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά στο ελέγξουμε Αρχιτή ψηφοφορία Πέρασε. Εγκρίθηκε λοιπόν το ψήφισμα. Επόμενη πρόταση ψηφίσματος. Ε, κατάσταση Μεσόγειο και ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ένωσης για τη Μετανάστευση της ΛΥΜΠΕ. Ε, το αρχικό κείμενο, παράγραφος 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, η τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Ε, στην παράγραφο 5 το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 στην παραγράφο 12 ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 12 η αρχική με ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ονομαστική κλίση. La Εγκρίνεται το αρχικό κείμενο. Μετά την αιτιολογική αναφορά 24, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2, υπέρ. Θέλετε έλεγχο. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Il Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 2 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η παριθμών 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη αιτιολογική σκέψη Β η τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται η έκθεση, το ψήφισμα. Grazie.